Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ, ώστε να ξεκινήσουμε τον οικονομικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων για την ετήσια έκθεση Ανάπτυξης και τα σχετικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τους ε, προσκεκλημένους μας, τον κύριο Ντομπρόσκης, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνο για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, τη Μαριάν Τάισεν, Επίτροπο Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κινητικότητας στο χώρο της εργασίας και τον Πιέρ Μοσκοβισή, Επίτροπο για Οικονομικές και Νομισματικών Υποθέσεις, ε, Φορολογία και Τελωνία. Καλώς ορίσατε σε αυτή την κοινή συνεδρίαση ε, Επιτροπής Απασχόλησης και Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, η οποία νομίζω ότι είναι μια σημαντική συνεδρίαση, διότι Σίγουρα η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση, διότι ξεκινά τον ετήσιο κύκλο της οικονομικής διακυβέρνησης, ε, το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά φέτος είναι πιο σημαντική όχι μόνο διότι συνεχίζονται οι δυσκολίες στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση της Ευρώπης, αλλά και γιατί είναι η πρώτη ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να έχει μια σαφή εικόνα και να είναι περισσότερο ε, έγγραφο οικονομικής στρατηγικής ε, παρά ε, απλώς και μόνο μία επισκόπηση και να βρίσκεται φυσικά στο επίκεντρο αυτό που αποκαλούμε μακροοικονομικό πακέτο, τη μακροοικονομική δέσμη μέτρων ώστε να υπάρχει και η κατάλληλη προβολή και συνεκτικότητα. Θα μας παρουσιαστεί λοιπόν η στρατηγική Υπάρχει και αυτό το ε, πρόγραμμα επενδύσεων, οι διαθερωτικές μεταρρυθμίσεις και ε, το θέμα της δημοσιονομικής ευθύνη, φιλικό ε, προς την ενέπτυξη βάσει της διαφοροποίησης και της προώθησης της εσωτερικής ζήτησης. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν υπάρχει και ο μηχανισμός επαγρύπνησης, ο alert mechanism, ε, για τη διαδικασία των μακροοικονομικών ισορροπιών, ο οποίος διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο, όπως επίσης και ε, το σχέδιο ε, της έκθεσης για τα θέματα αυτά. Είμαστε εδώ λοιπόν για να ακούσουμε τη νέα οικονομική ε, στρατηγική της Νέας Επιτροπής Juncker και να τη συζητήσουμε διότι θεωρούμε ότι και ανέκαθεν θεωρούσαμε άλλωστε και στο παρελθόν από τότε που ξεκίνησε η όλη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου Και επειδή ε, είμαστε περισσότερο επικεντρωμένοι πλέον στο νέο, οικονομικό στο ευρωπαϊκό εξάμεινο ε, και προσανατολιζόμαστε περισσότερο στην οικονομική πολιτική, είναι και ενισχυμένος ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο στην έκθεση Τάισεν, που φέρει πλέον το όνομα της Επιτρόπου μας, ζήτησε να υπάρχει και διοργανική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την ετήσια έκθεση ανάπτυξης και επομένως θεωρούμε ότι ήγηκε η ώρα να ξεκινήσουν συγκεκριμένες εργασίες επ' αυτού και με βάση και την μεγαλύτερη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα την αναφορά στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξη στην Κοινοβουλευτική Εβδομάδα. Θα γίνει φυσικά και φέτο και του χρόνου η Κοινοβουλευτική αυτή εβδομάδα και ε, ο οικονομικός αυτό διάλογος αποτελεί και μια ευκαιρία ε, για τους εισηγητές και τους κοιόδης εισηγητές για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να ξεκινήσουμε μια συζήτηση μαζί σας και φυσικά να υπάρχει και ένα έγγραφο το οποίο ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να επηρεάσει και τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου του Ευρωπαϊκού εξαμήνου στο Εαρινό Συμβούλιο. Αυτά είχα να σας πω εγώ και τώρα να δώσω απευθείας το λόγο στον πρώτο ομιλητή, στον κύριο Ντομπρόνσκης, Παρακαλώ κύριε Ντομπρόφσκης, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΚΟΝ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρώτα απ' όλα, εξ ονόματο Επιτροπή, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία να έχουμε αυτό τον κοινό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων με στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Απασχόλησης επίσης ως τμήμα της μακροοικονομικής διακυβέρνησης ε, και των διεργασιών και της εκκίνησης επίσης ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σήμερα λοιπόν η ομάδα μας, η Μαριάν και ε, εγώ θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα δέσμης μέτρων του 2015 και κάποια στοιχεία από αυτά έχουν ήδη παρουσιαστεί στο Ευρωκοινοβούλιο από τον πρόεδρο Γιούνκερ και τον αντιπρόεδρο Κατάινεν την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων για την Ευρώπη. Αυτή είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διευκόλυνση και ενδυνάμωση των επενδύσεων και αντανακλά επίσης μία από τις τρεις προτεραιότητες ε, για την ε, ετήσια ανασκόπηση για την ανάπτυξη για το 2015. Θα δώσουμε δηλαδή κίνητρα με αυτόν τον τρόπο στις επενδύσεις και θα συνεχίσουμε με τις διαθροτικές ε, μεταρρυθμίσεις και αλλαγές και την φορολογική υπευθυνότητα, δημοσιονομική υπευθυνότητα. Το 2015 λοιπόν η ε, ετήσια επισκόπηση ξεκινά ένα νέο κύκλο ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκού εξαμήνου θέτοντας ε, στόχους πολιτικής για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε την οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Θα έλεγα υπογραμμίζουμε με αυτόν τον τρόπο, τονίζουμε με αυτή την ιδέα και με τα έγγραφα που παρουσιάζουμε για το πώς θεωρούμε ότι ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο σαν αυτό πρέπει να διαμορφωθεί. Επίσης σημειώνουμε με ιδιαίτερη προσοχή την πρόσφατη έκθεση του κυρίου Ντεμπάκερ πώς μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω το ευρωπαϊκό εξάμεινο κάποιες ε, θετικές καλές ιδέες που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και να αναπτύξουμε. Και εν πάση περιπτώσει είναι επίσης η η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να εργαστούμε και να ενταχθεί έτσι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αποτελεσματικά σε αυτά τα πλαίσια και να ε, ενδυναμωθεί και να επιτηρηθεί εκ του σύνεγγης η δημοσιονομική διαδικασία και εξέλιξη και πώς μπορούμε από κοινού να διασφαλίσουμε ότι τα έντυπα, τα έγγραφα αυτά θα αποτελούν μέρος της κοινή μας στρατηγικής και θα εντάσσονται σε αυτήν για την ευδοκίμηση των στόχων μας για την ετήσια επισκόπηση και την έκθεσή μας, καθώς επίσης και είναι μια σαφής δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πράξει περισσότερα και να λάβει υπόψη περισσότερο κοινωνικούς δείκτες στο έργο το οποίο έχουμε ενώπιόν μας και νομίζω ότι η Μαριάν θα μπορέσει περαιτέρω να αναπτύξει αυτά τα σημεία είναι λοιπόν σημαντικό να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πρέπει να συνεργαστούμε και στο ευρωπαϊκό και στο εθνικό αλλά και στο περιφερειακό επίπεδο. Είναι κοινή η ευθύνη που έχουμε αναλάβει, έχουμε υπομειστεί αυτή. Και επίση πρέπει να συνεργαστούμε πολύ στενά εκ του σύνεγγυς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υλοποιηθεί, να επιτευχθεί αυτός ο στόχος που νομίζω ότι όλοι συμμεριζόμαστε και θέλουμε να ευδοκιμήσει για την ε, οικονομική ανάλυση αυτών των προτάσεων. Τι μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ξεπεράσει την ε, οικονομική και δημοσιονομική κρίση, όμως βλέπουμε δυστυχώς ότι είναι πολύ ευάλωτη η ανάκαμψη. Πρόσφατα στοιχεία για την ανεργία που έχουν δημοσιοποιηθεί από την ε, Eurostat καταδεικνύουν ότι βρίσκεται η ανεργία σε υψηλά επίπεδα και επίσης ή ε, αντιμετωπίζουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης ακόμα. Και σε σχέση με αυτό, με την κρίση, βλέπουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη ήταν πιο αδύναμη στην Ευρώπη από ό,τι σε μεγαλύτερες άλλες οικονομίες όπως την οικονομία των ΗΠΑ. Και αυτό πάλι αντανακλά θεωρούμε διαρθρωτικές αδυναμίες και ελλείψεις ε, της οικονομίας μας και όσον αφορά την αγορά εργασίας και την παραγωγή προϊόντων και παραγωγικότητα και βλέπουμε ότι οι επενδύσεις, οι επενδύσεις στην καινοτομία δεν επαρκούν πλήρως για να βελτιωθεί η παραγωγικότητα. Κατά την τελευταία δεκαετία αναπτύχθηκαν μη σώροπες σχέσεις ε, μακροοικονομικά στα κράτη της Ευρώπης και αυτό είναι ένας λόγος ε, που οδηγεί στο να παρεκκλίνουν και τα αίτια είναι η παρέκκληση των οικονομιών των κρατών μελών. Σε, σε κάποια κράτη-μέλη ενδυναμώνεται η οικονομία, όμως σε άλλα κράτη-μέλη παραμένει αδύναμη ακόμα. Και φυσικά δεν είναι όλα αποκλειστικά και μόνο κάποια νέα στοιχεία ή οι ειδήσει που απλά θα πρέπει μόνο να μας ε, ευαισθητοποιούν ή να μας ανησυχούν. Υπάρχουν όμως και θετικές ε, εξελίξεις και αυτό δείχνουν ε, οι οικονομικές προοπτικές από τις αναλύσεις μας. Αναμένουμε για πρώτη χρονιά οικονομική ανάπτυξη και στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά από του χρόνου. Και αυτό σίγουρα θα είναι μια θετική εξέλιξη. Καλά μαντάτα για πρώτη φορά ανάπτυξη, το τονίζω, και στα 28 συνολικά κράτη-μέλη και θα πρέπει έτσι να γίνουν αυτές οι προσπάθειες να ενισχυθεί αυτή η τάση, η προοπτική το 2016. Υπάρχει όμως ένα περιβάλλον χαμηλής ανάπτυξης, χαμηλού πληθωρισμού και υψηλής ανεργίας. Αυτό το μείγμα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί και πρέπει να είναι κύριο μέλημά μας να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση μέσω της μακροοικονομικής πολιτικής μας και διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα επενδύσεων λοιπόν είναι σίγουρα ένα από αυτά τα στοιχεία που όπως είπα πρέπει να συνοδεύεται επίσης εκ παραλίλου με διαθροτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Ταυτόχρονα όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε και τα θέματα ζήτησης και τα θέματα προσφοράς αμφωτέρωθεν δηλαδή και στις δύο πλευρές των οικονομικών αυτών παραμέτρων. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν σε σχέση με τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο βλέπουμε ότι την εμβάθυνση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς που πρέπει να ολοκληρωθεί με καλύτερη νομοθεσία και ρυθμίσεις Προχωρούμε λοιπόν, επίσης εργαζόμαστε και προχωρούμε με την ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά και αυτή είναι μια πρόσθετη ευκαιρία να σημειώσουμε ανάπτυξη, να σημειωθεί ανάπτυξη στην Ευρώπη και θα διοργανώσουμε, θέλουμε να διοργανώσουμε τα ενεργειακά σε μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση. Η κύρια λοιπόν ευθύνη για τις διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις εξακολουθεί να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Πολλά πρέπει να γίνουν σε σχέση με την αγορά εργασίας, με την παροχή υπηρεσιών και την ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών πολλά πρέπει να διοργανωθούν από τα κράτη-μέλη και να επιτευχθούν. Πρέπει να δημιουργηθούν τα, οι κατάλληλες προϋποθέσεις να υπάρξει ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και θα ακούσετε περισσότερα ευθύ στη συνέχεια επ' Δεύτερο, Δεύτερη παράμετρος, δημοσιονομική υπευθυνότητα. Τα προηγούμενα χρόνια χαρακτηρίστηκαν από την προσπάθεια δημοσιονομικής σταθερότητας. Εφέτος αλλά και του χρόνου αναμένουμε να υπάρξει μια αμερόληπτη ουδέτερη δημοσιονομικά διαμόρφωση των πραγμάτων. Η συνολική δηλαδή θέση δημοσιονομικά στα κράτη-μέλη θα είναι ουδέτερη δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει επιπρόσθετη λιτότητα, οι ούτε θα υπάρξει επι, ε, περαιτέρω κάποια αλλαγή. Υπάρχουν όμως κράτη-μέλη που επειδή εξακολουθούν να, να αντιμετωπίζουν ε, κάποια προβλήματα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τονώσουμε την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. εκεί. Επίσης για την παγίωση των εθνικών προϋπολογισμών ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να διευρύνουν τις επενδύσεις ε, και τις δαπάνες ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη και η φορολόγηση να ανακουφίσει τους εργαζόμενους την, ε, τον, την παράμετρο της εργασίας. Κάνοντας λόγο για τη μακροοικονομική διακυβέρνηση, επίσης ε, εργαζόμαστε σε ένα νέο πλαίσιο όσον αφορά την εξα, τις εξαπλές προτάσεις, six pack, την δέσμη μέτρων, την εξαπλή αλλά και την διπλή ε, που πρέπει να προχωρήσουν ε, όπως ε, σε μια νομισματική ένωση και παράλληλα με αυτά τα έγγραφα για τη μακροοικονομική διακυβέρνηση και τις προτάσεις μας είχαμε και την επισκόπηση των εξαπλών προτάσεων και των διτών προσπάθειων, six pack και two pack, θα ακούσετε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά μέσω στη συνέχεια. Όσον αφορά τώρα τα σχέδια προϋπολογισμών, δεν βρέθηκε κάποιο σχέδιο προϋπολογισμού που να παραβιάζει σε σημαντικό βαθμό ή να παρεκκλίνει σημαντικά από τις αρχές που έχουμε θέσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει καμία ένσταση. Φυσικά θεωρούμε ότι υπάρχει ένας αριθμός κρατών μελών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης ε, όσον αφορά τις ε, δράσεις ε, για την ανάπτυξη και βλέπουμε επίσης ιδιαίτερη επιβάρυνση λόγω του χρέους ε, σε ορισμένα κράτη. Σε αρκετά κράτη-μέλη παρακολύεται η ανάπτυξη από αυτή την επιβάρυνση της υπερχρέωσης. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε το έργο μας ε, για να συνεχιστεί η δημοσιονομική υπευθυνότητα και να διασφαλιστεί η αηφορία όσον αφορά την αντιμετώπιση της ε, κρατικής υπερχρέωσης των κρατικών χρεών. Τούτων λεχθέντων τώρα, στη συνέχεια και πάλι για άλλη μία φορά για την γενική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα κράτη-μέλη και τους εθνικούς προϋπολογισμούς, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει περισσότερο χρόνο στα κράτη-μέλη όσον αφορά την μη συμμόρφωση από πλευρά τους ε, με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά να ακολουθήσουν τις δεσμεύσεις τους ε, και να συμμορφωθούν, ιδιαίτερα για την Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο ισχύει αυτή η εξαίρεση, η παράταση. Είναι όμως σημαντικό αυτά τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν εκ του σύνεγγυς αυτές τις υποχρεώσεις, να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις και φυσικά σε σχέση με τη μακροοικονομική διακυβέρνηση για τις διάφορες αποφάσεις και δυνατότητες που θα έχουν να δράσουν όπως πρέπει. Θα ήθελα να ολοκληρώσω υπογραμμίζοντας ότι η κύρια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι να διευκολυνθεί η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται και θα διατηρείται η νομισματική σταθερότητα. Και γι' αυτό προσβλέπουμε και αδειμονούμε να υπάρξει μια θετική συνεργασία μεταξύ μας και μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα πρέπει να συνεχιστεί η πίεση ώστε όσον αφορά το ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο να προχωρήσουμε εναρμονισμένα και ε, εκ παραλίλου όλοι, ώστε να υπάρξει αηφορία για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε Ντομπρόσκης, και τον να το λόγο στην Επίτροπο Τέισεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιας και έχω η ερμηνεία στη διάθεσή μου, θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα. Πρόεδρε, συνάδελφοι. Καλοί συνάδελφοι, οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά από την παρουσίαση του Αντιπροέδρου Ντομπρόφσκης θα επισέλθω σε λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά ε, τα θέματα απασχόλησης ε, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Η επιτυχία των οικονομικών φιλοδοξιών μας έχει να κάνει ε, με την υγιή ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής ε, αξιοπιστίας και φιλοδοξής ε, επένδυσης. Θα πρέπει λοιπόν οι διαθετικές επενδύσεις να πραγματοποιηθούν και κυρίως σε αυτή την τρίτη πτυχή θα επικεντρωθώ μαζί με τα άλλα έγγραφα που παρουσιάστηκαν. Υπάρχει και η έκθεση για το σχέδιο έκθεσης για την απασχόληση. Και αυτό καταδεικνύει με μεγάλη σαφήνεια ότι είναι απαραίτητο να γίνουν μεγάλες ε, μεταρρυθμίσεις γιατί υπάρχουν ε, μεγάλα προβλήματα, αν και έχει σημειωθεί κάποια μικρή πρόοδο στα θέματα απασχόλησης. κοιτώντα το συνολικό ποσοστό ανεργίας, έχει βελτιωθεί από 10,8% σε 10,1% σε ένα χρόνο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα 24,6 εκατομμύρια ανέργους, 10,1% του πληθυσμού όπως σας είπα. Και αν κοιτάξουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα στοιχεία αυτή, διαπιστώνουμε ότι είναι εξαιρετικά υψηλή ενεργεία μεταξύ των ε, νέων. 1,9% ήταν η βελτίωση σε ένα έτος. Ορατή η βελτίωση, αλλά και πάλι το 21,6% ως ποσοστό ανεργία των νέων είναι κάτι απαράδεκτο και η μακροπρόθεσμη ανεργία είναι μεγάλο πρόβλημα. Το ίμιση των ανέργων είναι μακροπρόθεσμα ανέργη. Πάνω από 12 εκατομμύρια άνθρωποι δηλαδή. Και η ανισότητα στα εισοδήματα και η φτώχεια έχουν αυξηθεί σε πολλά κράτη-μέλη σε σύγκριση με την αρχή της κρίσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ έχουμε αποτύχει σε ό,τι αφορά τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2020. Αντί να έχουμε μειώσει τους στόχους κατά 20 εκατομμύρια, έχουν αυξηθεί κατά 6 εκατομμύρια. Φυσικά έχουν καταβληθεί προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, καλές προσπάθειες και βλέπουμε ότι οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς, αλλά αυτό που δεν επιτρέπεται να κάνουμε είναι να τελματώσουμε και να θεωρήσουμε ότι από μόνο τα πράγματα θα κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ζητώ λοιπόν την υποστηρίξή σας σε ό,τι αφορά την πρόκληση αυτή που αφορά την ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πρέπει ασφαλώς να συνεχίσετε να διασφαλίζετε στο μέλλον. Και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εστιάζεται σε πέντε σαφείς προτεραιότητες. Καταρχάς, θέλουμε να δημιουργηθεί θέσεις απασχόλησης και να υποστηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, να υποστηρίξουμε τη δημιουργία θέσεων εργασία μέσω του επενδυτικού προγράμματο το οποίο εκκινήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλουμε ο κατακαιρματισμό τη αγορά εργασία να αντιμετωπιστεί και η καταπολέμηση της ε, μαύρης εργασίας. Επίσης να υποστηριχθεί Επίσης ε, η επιβάρυνση της εργασίας θα πρέπει να μετατοπιστεί σε άλλο τομέα που δεν θα επιβαρύνει την δημιουργία θέσεων εργασίας. Κατά τέταρτον, να επενδύσουμε σε επαγγελματικά προσόντα και εκπαίδευση προκειμένου οι νέοι να έχουν τις βέλτιστες δυνατές δυνατότητες και ικανότητες ε, στο μέλλον και να εξυγχρονίσουμε τους μηχανισμούς προστασίας προκειμένου και τα παιδιά μας να μπορούν στο μέλλον να επωφεληθούν. Θα ήθελα να πω ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν εστιάζονται μόνο στην απασχόληση και στην κοινωνική προστασία. Δεν γίνεται να εστιάζονται μόνο σε αυτούς τους κλάδους. Αν θέλουμε μεγαλύτερη απασχόληση και πιο μεγάλη συνοχή στην κοινωνία, θα πρέπει να στραφούμε και άλλους, σε άλλους τομείς, στα προϊόντα, στις ε, υπηρεσίες, στην καινοτομία, στην ποιότητα των κρατικών υπηρεσιών και για αυτό το λόγο το επενδυτικό μας πρόγραμμα, το οποίο και ακούσατε πριν από λίγο, περιλαμβάνει και ε, εμπόδια για συγκεκριμένες επενδύσεις, τις οποίες δεν θέλουμε να ανεχτούμε. Αυτά λοιπόν θα θέλαμε να τα ενθαρρύνουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών μέσω ενός ε, ισχυρού κοινωνικού διαλόγου προκειμένου όλοι στην κοινωνία να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Με την Επιτροπή λοιπόν, ε, στα πλαίσια της Επιτροπής συναντηθήκαμε με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και θέλουμε αυτή η συνεργασία να συνεχίσει να διαμορφώνονται με στεναρό τρόπο. Μαζί με τους εταίρους μας λοιπόν εξετάζουμε πώς τους επόμενους μήνες μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε και πώς μπορούμε να αναλάβουμε μια εντυπωσιακή τέτοια πρωτοβουλία. Αγαπητοί βουλευτές, να έχουμε υπόψη μας ότι η ανεργία και συγκεκριμένα η μακροπρόθεσμη ανεργία και η ανεργία των νέων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η οικονομία μας. Η ανεργία και η μεγάλη φτώχεια αποτελούν μακροοικονομικές ανισότητες που αποσταθεροποιούν την κοινωνία μας και γι' αυτό λοιπόν σήμερα ξεκινήσαμε την αναβάθμιση των κοινωνικών δικτών και των δικτών απασχόλησης στη διαδικασία τη μακροοικονομική του επόμενου έτους. Ο συνάδελφος Μοσκοβισή ενδεχομένως να αναφερθεί στα συντήματα αυτά, αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι στη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε κάποιους κοινωνικούς δείκτες, προκειμένου και αυτοί να ληφθούν υπόψη κατά την ε, εις ανάλυση της κατάστασης ανακρατος μέλος, προκειμένου να έχουμε και μια καλή επισκόπηση της κοινωνικής κατάστασης στα κρατημέλη. Και έτσι να μπορούμε ίσως να αντιδρούμε πιο γρήγορα, πιο σωστά, πιο έγκυρα στις κοινωνικές προκλήσεις της Ευρώπης και χαίρομαι που και στον τομέα αυτό έχει σημειωθεί καλή πρόοδος και ελπίζουμε να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Με τη δική σας υποστήριξη, αγαπητοί βουλευτές, θα ήθελα να συνεχίσω να εργάζομαι προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, την ε, κυρία Τέισεν. Και τώρα είναι η σειρά του Πιέρ Μοσκοβισή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Θα μιλήσω αργότερα στη διάρκεια της ημέρας για τα προσχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα αυτά, αλλά τώρα θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την έκθεση για το μηχανισμό επαγρύπρησης, ε, την οποία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη Παρασκευή μαζί με την δέσμη οικονομικών μέτρων που ανέφερε ο Πρόεδρος στα πλαίσια της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης που ανέφερε ο συνάδελφος Ντομπρόσκης. Θα σας παρουσιάσω εντάχει λοιπόν τα στοιχεία της έκθεσης και το τι ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε για το πρώτο εξάμεινο του 2015. Καταρχάς να σας υπενθυμίσω ότι η έκθεση αυτή είναι το σημείο κίνησης του ετήσιου κύκλου για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και στόχος είναι είναι να εντοπίσουμε και να ρυθμίσουμε τις ελλείψεις ισορροπίες οι οποίες ε, ε, δημιουργούν πρόβλημα στην αγαστή λειτουργία της οικονομίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσε φυσικά να υποσκάψει και την ε, καλή λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Στην έκθεση εντοπίζονται τα κράτη-μέλη τα οποία θα μπορούσαν να πληγούν από τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα οικονομικής πολιτικής και γι' αυτό ακριβώς στα κράτη αυτά θα γίνει μια εις βάθος εξέταση. Ε, η έκθεση για, την, ε, ε, το μηχανισμό επαγρύπνησης περιλαμβάνει κάποια αρχική αξιολόγηση και μόνο μετά την εισβάθος ανάλυση θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει στο συμπέρασμα για το κατά πόσον υπάρχουν ανισορροπίες ή κάποια υπερβολικά ελλείμματα πλεονάσματα. Φέτος έχουμε 16 κράτη-μέλη που επιλέγησαν για επιπλέον ανάλυση. Από αυτά τα 14 ε, επιλέγησαν με βάση την εις εξέταση που έγινε την προηγούμενη χρονιά. Στην περίπτωση της Κροατίας, της Ιταλίας και της Σλοβενίας ε, θα εξεταστεί κατά πόσον οι υπερβολικές ανισορροπίες που διαπιστώθηκαν στο παρελθόν ε, αμβλήνονται, επιμένουν ή επιτείνονται και αυτό φυσικά θα πρέπει να Εκύψει και με συνεισφορά των κρατών μελών για να διορθωθούν αυτέ οι ανισορροπίε. Για την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ουγγαρία είναι χώρε οι οποίε χρειάζονται κάποια αποφασιστικά μέτρα. Η αξιολόγηση θα ε, δει κατά πόσον υπάρχουν κίνδυνοι που ε, σχετίζονται με την επιμονή αυτών των, ε, τη συνέχιση αυτών των ανισορροπιών. Και όσον αφορά τα κράτη-μέλη τα οποία διαπιστώθηκε στο παρελθόν ότι υπήρχε ανισορροπίες, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γερμανία, κάτω χώρες, η Φιλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, θα ε, εξετάσουμε κατά πόσον σε κάποιες από αυτές τις χώρες ε, συνεχίζονται οι ανισορροπίες και θα πρέπει να διορθωθούν. Αυτά λοιπόν για τις 14 χώρες που είχαμε στο παρελθόν. Για πρώτη φορά τώρα θα γίνει και ε, περαιτέρω εξέταση και για την Πορτογαλία και για τη Ρουμανία. Η Πορτογαλία ε, κατάφερε να εφαρμόσει το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής ε, στο μέσα του 2014 και ανήκει πλέον στις χώρες που βρίσκονται ε, στη διαδικασία της συνήθους Αυτά λοιπόν ω απολογισμό τη κατάστασης. Τώρα να περάσουμε στην ει εξέταση των οριζόντιων εξελίξεων που έχουμε στην έκθεση. Τα οριζόντια θέματα αφαινούν καταρχάς ε, την εξωτερική ε, αποκατάσταση της ισορροπίας. Ε, υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες είναι υπερχρωμένες που έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ σημαντική συσσόρευση χρέους παρά το γεγονός ότι έχουν μειώσει ουσιαστικά τα ελλείμματά τους. Υπάρχει επίσης και μια ασύμετρη κατάσταση με χώρες οι οποίες είναι καθαροί πιστωτές ε, και υπάρχουν ε, ε, συνεχή πλεονάσματα εκεί και επομένως αυτό μπορεί να αποδυναμώσει τη ζήτηση και τις επενδύσεις. Επίσης εξετάζουμε τι γίνεται με την ανταγωνιστικότητα. Ε, περισσότερο προς τη σωστή κατεύθυνση για αρκετές χώρες εδώ. Διαπιστώνουμε επίσης ότι υπάρχει μια ετερεγένεια στη διαδικασία της ε, αποπληρωμής του χρέους, ε, διότι υπάρχει ακόμα πολύ ψηλό χρέος για τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτή η ετερογένεια φυσικά σχετίζεται και με τις διαφορές που έχουμε στον πληθωρισμό και την αύξηση του ΕΠ. Εξετάζουμε επίσης και την ετερογένεια στο σεβαστικό τομέα. Ε, εξετάζουμε την κατάσταση του τραπεζικού συστήματος επιπλέον. Ε, υπάρχουν κάποιες αλλαγές και υπάρχουν ε, αποτελέσματα της ε, ετήσιας έκθεσης ε, ποιότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δείχνουν ότι σε γενικές γραμμές έχουν μειωθεί η κίνηση. Ε, βλέπουμε επίσης και την ισχνή ανάπτυξη της πίστοσης. Αυτό λόγω της προσφοράς καταρχάς, αυτό σχετίζεται με την υπερχρέωση ε, κάποιων χωρών και φυσικά και τη ζήτηση των πιστώσεων που σημαίνει ότι δεν έχουμε πολύ καλές επενδύσεις. Ε, η συνάδελφος Τέισαν αναφέρθηκε και στη σχέση με την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα και συμφωνώ μαζί της ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιοι νέοι κοινωνικοί δείκτες ε, και τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Λάβαμε υπόψη, υπόψη μας ούτως ή άλλως τους κοινωνικούς δείκτες για να καταλάβουμε καλύτερα τι δυνατότητες έχουμε για νέα κατανομή πόρων και προσαρμογή στις δυνατότητες παραγωγής της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά θα τα δούμε ε, στην εισβάθος ανάλυση ούτως ή που θα κάνουμε στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Συμφωνώ επίσης ε, με την Μαριάνο ότι η κοινωνική διάσταση ε, είναι ουσιαστικό στοιχείο της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπαθούμε να την ενισχύσουμε. Ολοκληρώνοντας κύριε Πρόεδρε, θα να σας πω ότι αυτά όλα θα συζητηθούν και στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ και λογικά θα πρέπει να εγκρίνει επισήμως και τα συμπεράσματα όλων αυτών. Ε, εν αναμονή αυτών θα ήθελα να δω και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά ε, και φυσικά βάσει των συζητήσεων μεταξύ του Συμβουλίου και της ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Eurogroup φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ετοιμάσει μια έκθεση για το Μάρτιο του 2015 ε, και εκεί ε, θα δούμε και τις συστάσεις αναχώρησης χώρα, τις ε, Country Specific Recommendation και θα έχουμε και κάποιες ουσιαστικές αποφάσεις ε, σε περίπτωση που υπάρχουν υπερβολικά ελλείμματα και θα, όλα αυτά θα ε, αποφασιστούν με βάση τον απολογισμό που θα κάνουμε το Μάρτιο. Αυτά κύριε Πρόεδρε για το μηχανισμό επαγρύπνησης. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ τον Πιέρ Μοσκοβισή και τους υπόλοιπους ε, επιτρόπους και τώρα να περάσουμε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στους δύο εισηγητές ε, στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και Επιτροπή Απασχόλησης ε, για τρία λεπτά στον καθένα και θα έχουμε οκτώ λεπτά σύνολο για τις απαντήσεις των Επιτρόπων. Ο Ντάριος Ροζάτη έχει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τρεις επιτρόπους για τις παρουσιάσεις τους. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ σημαντική χρονική συγκυρία σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, στην αρχή της διαδικασίας λοιπόν το 2015 και νομίζω ότι η όλη άσκηση θα καθορίσει τις προσπάθειες και τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν του χρόνου για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασία στην Ένωση. Δύο ερωτήσει έχω να απευθύνω προ του προσκεκλημένου μα σήμερα. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει σε ότι τα θέματα που αφορούν την ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων. Η ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων. Επενδυτικό ε, κομμάτι, κομμάτι δημοσιονομικής πειθαρχία και το κομμάτι των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Τα ποσοστά των τριών αυτών πυλώνων, λοιπόν, ποια πιστεύετε ότι είναι η σωστή ισορροπία μεταξύ των τριών και ποια είναι η πρόοδος που έχει σημειωθεί μεταξύ των τριών αυτών πυλώνων, που, που έχουμε την λιγότερη πρόοδο και ποια είναι η σχέση μεταξύ των μακροοικονομικών εξελίξεων σε κάθε χώρα και των τριών αυτών μετόπων. Υπάρχει σχέση πιο συγκεκριμένα μεταξύ της αργής ε, εξέλιξης των διευθυντικών μεταρρύθμισεων σε χώρες όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανισορροπιών και σοβαρά θέματα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς δείκτες, ε, πέρα από το scoreboard, ποια είναι η διαδικασία λοιπόν χρήσης των κοινωνικών δικτών σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της αξιολόγησης στα πλαίσια του μηχανισμού αξιολόγησης και ενδεχομένω και στην εις ανάλυση σε αντίθεση με τους οικονομικούς δείκτες όπου έχουμε σαφή κατόφλια, σαφείς ορισμούς, έχει οριστεί η διαδικασία σε ποιο βαθμό όμως οι κοινωνικοί δείκτες ε, θα επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και σε ποιο βαθμό είναι απλά μια πηγή καλύτερης κατανόησης της μακροοικονομικής κατάστασης. Σας ευχαριστώ. Επόμενος μιλητής, ο Σέρτζιο Γκουτιέρες Πιέτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ επίσης την κοινή αυτή εμφάνιση των τριών επιτρόπων εδώ ενώπιον μας στην έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου γιατί συσχετίζονται οι αρμοδιότητες τους. Οι βαθιές αλλαγές σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν από τον κύριο Ντομπρόφσκι και τον κύριο Μοσκοβίση και αυτά που μπορούν να, να γίνουν και από την κυρία Τάισεν θα είναι θεραπευτικές δράσεις. Ε, αν δεν αλλάξουν ε, οι πολιτικές ε, δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σχέση με την απασχόληση θέματα που αναφέρθηκαν προηγούμενα. Αληθεύει ότι καλά ακούγονται αυτά σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο σε σχέση με την αλλαγή, αέναρξη αλλαγή όσον αφορά την μακροοικονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε, είναι, είναι Πώ φιλόδοξες αυτές οι αλλαγές για να προαχθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, διαφορετικές θέσεις απασχόλησης από το ότι έγινε μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό πρέπει να διατυπωθούν ερωτήματα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν εμφαίνονται σε αυτή την ε, επισκόπηση. Ο μεγάλος κίνδυνος που σήμερα έχουμε υπό το πρίσμα των ανισορροπιών μακροοικονομικά και για την απασχόληση το επίπεδο μακροχρόνια ανέργων για παράδειγμα που είναι ανησυχητικό καθώς επίσης και επάρκεια μισθού για να μπορέσει να ξεφύγει ο εργαζόμενος από την παγίδα της φτώχειας δεν εμφαίνονται ούτε και οι παρεκκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ αυτών των παρεκκλήσεων με μεγάλες ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών και αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος μακροοικονομικά. Επίσης για την δημοσιονομική ευθύνη σε σχέση με τις ε, πολιτικές που ακολουθήθηκαν χρησιμοποιούνται όλα τα περιθώρια τα οποία προβλέπονται από την, ε, το, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ώστε να είμαστε πιστοί με την, ε, για την οικονομική ανάπτυξη και για αυτούς τους λόγους πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε περισσότερο υπόψη ότι η μεγάλη έλλειψη που υπήρχε κατά το παρελθόν ήταν ότι δεν υπήρχε συντονισμός ε, και αναλογία σε σχέση με τις δράσεις για τη μείωση του χρέους ε, και των προβλέψεων της οικονομικής ανάπτυξης που γινόντουσαν από τα κράτη-μέλη. Συμμετέχω για τρίτη φορά σε αυτή τη συζήτηση και πάντα από τον αρμόδιο επίτροπο για το οικονομικό τμήμα άκουγα ότι θα έχουμε ανάπτυξη πάνω από ένα λέει 100. Κάθε φορά που γινόντουσαν τέτοιες προβλέψεις, τις τελευταίες φορές ε, έχασαν όλες το στόχο τους. Δεν υλοποιήθηκαν. Γι' αυτό λοιπόν, ναι μεν σύμφωνο ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν διαθωτικές αλλαγές για την ανταγωνιστικότητα. Όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις για την αναζήτηση της ανταγωνιστικότητας ε, όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ή των των ενεργειακών αγορών ε, με την μισθολογική υποβάθμιση που υπήρξε που ήταν τεράστια σε πολύ μεγάλη εμβέλεια δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερώτηση λοιπόν, είναι πρόθυμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα αναγνωρίσει αυτά. Διότι για παράδειγμα διαβάζω σε αυτή την επισκόψη ανάπτυξη ότι υπάρχει θετική λέει αναγνώριση για τις ε, ε, επανορθώσεις που έγιναν. Δεν λαμβάνεται όμως υπόψη σε κάποιες χώρες υπήρξε μισθολογική υποβάθμιση των χαμηλών χαμηλότερων μισθών πάνω από 15% πράγμα το οποίο δημιουργεί τεράστια ανισότητα. Θα επανορθώσει αυτές τις ανισότητες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ελάχιστων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρξει ασφάλιση κατά της ανεργίας. Είναι πρόθυμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υλοποιήσει αυτές τις δεσμεύσεις ώστε να υλοποιηθούν οι φιλοδοξίες. Ευχαριστώ. Οκτώ λεπτά και οι τρεις έχετε να απαντήσετε από την Επιτροπή. Πρώτος ο Βάλτης Ντομπρόσκης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και ξεκινώ με τις ερωτήσεις του κυρίου Ρωσάτη. Πρώτον, για την ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων. Θα έλεγα και οι τρεις πυλώνες είναι πολύ σημαντικοί και δεν έχουμε κάποια αναλογία που να έχουμε επιμερίσει σε κάθε πυλώνα ξεχωριστά. Και αυτό επειδή θεωρούμε ότι όλοι και οι τρεις αυτοί πυλώνες συνεμπλέκονται και έχουν την αναλογία τους στην εξίσωση αυτή μεταξύ των τριών. Για το θέμα πόσο ενεργά θα εργαστούμε ώστε να υπάρξει η επιμερισμένη η ισότιμη εμπλοκή των τριών πυλώνων έχουμε το πρόγραμμα της ε, επένδυσης ε, ε, που προβλέπονται δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την τόνωση των δραστηριοτήτων στην Ευρώπη από πλευράς επιχειρήσεων θα διευκολυνθούν λοιπόν οι ιδιωτικές επενδύσεις όχι μόνο με το μέσο αυτού του σχεδίου, αυτού του προγράμματος αλλά θα υπάρξουν και δημόσια κονδύλια για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Αλλά επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν οι πιο θετικές ε, προϋποθέσεις για να ε, ευδοκιμήσει η προσπάθεια του ιδιωτικού τομέα. Στη συνέχεια διαθεωτικές μεταρρυθμίσεις. Ε, σημαντικό αυτό το έργο και πρέπει να συνεχιστεί. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω αυτής της δράσης να διασφαλίσουμε την αηφορία στην οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σίγουρα αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική παράμετρος ε, ε στη συνέχεια δημοσιονομική υπευθυνότητα. Αναμένουμε να μπορέσει να προαχθεί και φέτος ε, και του χρόνου και είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε με αυτόν τον υπεύθυνο τρόπο την πορεία μας. Να μην δημιουργηθεί μια νέα, εκ νέου κρίση εμπιστοσύνης όπως ε, την ζήσαμε, την βιώσαμε πριν από πέντε χρόνια για παράδειγμα. Και να, γιατί αυτό θα έχει σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις δεν μπορούμε με κανένα τρόπο λοιπόν να αμελήσουμε τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις και την ε, ε, <clears throat> δυνατότητα της ε, δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Το έργο αυτό, όπως ε, προαναφέρθηκε, έχει ξεκινήσει για να ενισχυθεί και η κοινωνική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια σε βάθος ανάλυση για την ε, ε, απασχόληση χρησιμοποιούνται δείκτες ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες. Θα το επαφήσω στην κυρία Τάισεν να αναπτύξει περισσότερο αυτό το θέμα αυτών των δικτών που προάγουμε εμείς ε, ε, με ιδιαίτερο τρόπο. Και για τις ερωτήσεις ε, του επόμενου Ευρωβουλευτή που ήταν αρκετές, πρώτον αν αυτά τα σχέδια, τα προγράμματα είναι αρκετά φιλόδοξα ρώτησε. Θα έλεγα αυτό το οποίο εμφανίζεται στην ετήσια επισκόψη για την ανάπτυξη το μέσω της δέσμης μέτρων μακροοικονομικών, ε, μακροοικονομικής πολιτικής είναι τα πρώτα βήματα που χρειάζονται και πρέπει να γίνουν και χρειάζεται να γίνουν και πρέπει η ζήτηση και η προσφορά στην οικονομία να συνεξεταστούν και όλα τα τρία στοιχεία τα οποία ε, ε, εμφαίνονται και παρουσιάζονται να αλληλοσυμπληρούνται και να έχουν παραπληρωματική λειτουργία για την επίτευξη των στόχων. Και στη συνέχεια για κάποια ερωτήματα που αναφέρατε για την ε, ελαστικότητα, την ευληγησία αυτό είναι κάτι που ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας απασχολεί και κατά την έναρξη του επόμενου έτους, ε, αρκετά νωρίς δηλαδή, θα έχουμε μια ανακοίνωση που θα εκδώσουμε για την ε, καλύτερη δυνατότητα της χρήσης του μέσου ελαστικότητας και όσον αφορά ελάχιστους μισθούς, αυτό είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει να προαγάγουν τα κράτη-μέλη ώστε να βρίσκονται σε αντιστήχηση και αναλογία σε σχέση με την παραγωγικότητα των κρατών μελών ή μισθή και σε σχέση με την ε, δυνατότητα αυτή πρέπει να συνεχιστεί από τα κράτη-μέλη σε σχέση με τους ελάχιστους μισθούς. Ευχαριστώ. Μαριάν Τάισεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική και τις θέσεις απασχόλησης. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω αυτό που κατέστη σαφές ότι ακόμα και στην ίδια την ερώτηση των βουλευτών έγινε σαφές αυτό, ότι αν θέλουμε ε, να βελτιώσουμε και να υποστηρίξουμε την απασχόληση θα πρέπει να βασιστούμε στην προσφορά και στη ζήτηση και θα πρέπει να κοιτάξουμε τις επενδύσεις ε, να υπάρξουν και πάλι επενδύσεις, να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις για να υπάρξει καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερα προσόντα. Προσόντα λοιπόν, επαγγελματικές ικανότητες, αυτή είναι η λέξη κλειδί και θα πρέπει να δούμε και την κοινωνική μας προστασία. Θα πρέπει να προστατεύει αλλά και να δραστηριοποιεί η κοινωνική προστασία σε ό,τι αφορά τους κατώτατους μισθούς που ρωτήσατε. Όπως ε, είπε και ο συνάδελφός, είναι κάτι που θεωρούμε ότι είναι καλό να υπάρχει ένα κατόφλι, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να υποβάλει προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Απλά, λοιπόν, ενθαρρύνουμε τα κρατημέλη, αλλά δεν μπορούμε να τα υποχρεώσουμε σε ό,τι αφορά τους κατώτατους μισθούς και θα θέλαμε να δημοσιεύσουμε ε, προτάσεις για ε, μισθούς αναφοράς, αλλά κάθε χώρα ε, λοιπόν έχει δική της αρμοδιότητα. Μόνο να ενθαρρύνουμε μπορούμε από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς δείκτες τελευταίο σημείο. Εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή προκειμένου να ενταχθούν καλύτερα στο πλαίσιο των μακροοικονομικών ανισοτήτων, ανισορροπιών. Ήδη συμβαίνει αυτό σε ό,τι αφορά την ε, έκθεση ετήσιας ε, ανάπτυξης, θα δείτε ότι υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση στα θέματα κοινωνικής ανάπτυξης. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό δικτών και να θέσουμε κατόφλια. Και αυτό λοιπόν ε, θα το κάνουμε μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα το κάνουμε μόνοι μας, αλλά σίγουρα πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Και τα πιο σημαντικά θα είναι σίγουρα τα κατόφυλλα που θα έχουν να κάνουν με το βαθμό ε, δραστηριότητας και ανεργίας. Όπως σας είπα, η φτώχεια και η ανισότητα στην κοινωνία είναι σημαντικοί παράγοντες, αλλά κοιτώντας στις αναλύσεις της ανισότητας και της φτώχειας, βλέπουμε ότι αυτά έχουν να κάνουν σχεδόν εξ ολοκληρού με την ανεργία. Όποιος δεν δουλεύει βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να δραστηριοποιηθεί ο κόσμος. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης της ε, φτώχειας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μοσκοβισή. Πολύ σύντομα για να συμπληρώσω αυτά που είπε ο Βαλτής και με τα οποία συμφωνώ πολύ του. Η ισορροπία μεταξύ των τριών πυλώνων. Δεν μπορούμε να προτιμήσουμε τη μία υπέρ της άλλης τον έναν μάλλον υπέρ των άλλων. Υπάρχει όμως έναν που είναι ε, πιο ε, καινούριο ε, και είναι ο πυλώνας των επενδύσεων. Επομένως θα πρέπει να δούμε τι προκλήσεις έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή με τους Ευρωπαίους, την ισχνή ανάπτυξη, ε, ισχνό πληθωρισμό και ε, αυξημένη ενεργεία. Κάτι το οποίο είναι και από πολιτικής και από κοινωνικής ε, σκοπιάς απαράδεκτο. Και επομένως θα πρέπει να δούμε ποια είναι το βασικό στοιχείο του ελλείμματος και της ανάπτυξης και αυτό είναι το ποσοστό των επενδύσεων. Αν δούμε το ποσοστό των επενδύσεων των Ευρωπαίων σε σχέση με το τι συνέβαινε το 2008, διαπιστώνουμε ότι σήμερα κάθε χρόνο είμαστε 20% κάτω στις επενδύσεις σε σχέση με το 2008. Και αυτό φυσικά είναι πολύ σημαντικό, διότι μπορεί να οδηγήσει σε ε, απόσταση μεταξύ των σημαντικότερων ανταγωνιστών μας και κυρίως με τη ΣΥΠΑ. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να ανακάμψουμε, να βελτιώσουμε αυτές τις απώλειες, να διατηρώσουμε ε, τις διαρθρωτικές αλλαγές και να προσθέσουμε και αυτό τον πυλώνα των επενδύσεων με ένα ρυθμό τον οποίο ε, θα μας επιτρέψει να δημιουργήσει με αυτή τη συνοχή στην οποία αναφέρθηκε ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη στην εισαγωγή του. Και να πω, και εδώ έχουμε ένα δεύτερο στοιχείο, ότι υπάρχει ένας νέος κύκλος ο οποίος ανοίγεται αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα οι Ευρωπαίοι ήταν σε ένα στάδιο σταθεροποίησης μετά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Ό,τι κάναμε, ο καθορισμός του προγράμματος προσαρμογής, η Τραπεζική Ένωση, όλα όσα ε, πήγαν προς την κατεύθυνση της επίλυσης της τάδε τη δίνα κρίσης και η δημιουργία του μηχανισμού σταθερότητας, ε, μας οδήγησαν πλέον σε μια νέα φάση. Έχουμε πλέον σταθερότητα, αλλά τώρα πρέπει να υπάρξει μια ε, δυναμική και μια κίνηση. Ο ε, συνάδελφος Ντομπρόσκης είπε ότι υπάρχει διάθεση να χρησιμοποιήσουμε το σύνολο των μηχανισμών που έχουμε στη διάθεσή μας και να δράσουμε στο πλαίσιο των ε, υφιστάμενων ε, εργαλείων. Σίγουρα δεν έχουμε χρησιμοποιηθεί επαρκώς, αλλά και με την ευελιξία που μας επιτρέπεται. Θα παρουσιάσουμε και μία ανακοίνωση στις αρχές του επιμένου έτους στην ευελιξία στα πλαίσια των κανόνων ε, οι πρώτες ε, ε, ενδείξεις υπάρχουν ήδη στην παρουσίαση του σχεδίου επενδύσεων του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του κ. Γιούνκερ και του Γιούργη Κατάινεν για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το κεφάλαιο του στρατηγικού ταμείου επενδύσεων που θα δημιουργηθεί και φυσικά να μπορέσουμε να έχουμε και τις κατάλληλες επενδύσεις. Ευχαριστώ να δώσω τώρα τα ενία της ε, Προεδρίας ε, στη συνάδελφο τη Μαρίτα Ούλσφορ και να υπενθυμίσω σε όλους εσάς ότι για να μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο θα πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από όλους να είναι σύντομοι και επίσης από τους επιτρόπους ε, να κάνουν κατάλληλη κατανομή του χρόνου που τους διαθέτουμε, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά το χρόνο μας. Να διαβάσω τον κατάλογο των ομιλητών. Ε, ε, Μονό, Σογκόρ, Σάντερ. Μαρίζα, Μαρίζα, παρακαλώ. Κυρία Φρέιρα. Α, να ξεκινήσουμε λοιπόν με το δεύτερο γύρο μιλητών. 1,5 λεπτό για κάθε έναν από τους κοιόδης συζητητές, 10 λεπτά συνολικά για τους επιτρόπους για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Και να ξεκινήσουμε με τον ε, κύριο Σάντς από την ομάδα των σοσιαλιστών από την ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, η μεγάλο ποσοστό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την εθνική αγορά ε, τροφοδοτούνται και δεν ε, ευνοούνται μακροπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα από την ε, ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα. Όμως πρέπει να γίνει αυτό. Η ε, παγίωση και εξυγίανση δημοσιονομικά θα πρέπει να μπορέσει να δώσει την δυνατότητα στα κράτη ώστε να δώσουν τα κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεν είναι αυτή η κατάσταση η οποία όμως ε, διακηρύσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση με τα όσα γίνονται. Ευχαριστώ. Sofia Ribeiro from EPP. Η Σοφία Ριμπέρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Οι προκλήσεις που τίθενται είναι να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των προτεραιοτήτων κοινωνικών και οικονομικών που αλληλοσυνδέονται να δούμε την κατάσταση μεταξύ των ε, κρατών μελών και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ε, από πλευρά ε, του ΕΛΚ χαιρετίζουμε την νέα αυτή προσπάθεια για την δημοσιονομική ανάπτυξη κίνητρα για τις, για τις επενδύσεις που πρέπει στους πυλώνες αυτές, αυτούς να εντάσσονται και να υπάρξει η αντιμετώπιση της υπερχρέωσης. Προγράμματα για τις υποδομές, ενεργειακές υποδομές, υποδομές στην εκπαίδευση εκπαίδευση, κατάρτιση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αποδοτικότητα της ε, εκμετάλλευσης ενέργειας. Πρέπει να υπάρξει η ποιότητα δημοσιονομικά για τη δημιουργία μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς που θα συνδυάζει την ελευθερία της αγοράς με την δικαιοσύνη, την κοινωνική δικαιοσύνη. Πρέπει να δημιουργηθούν εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης στα επόμενα χρόνια. Είναι ένας φιλόδοξος στόχος αλλά ανεπαρκής ε, για να αντιμετωπιστούν τα σχεδόν 25 ε, εκατομμύρια ανέργων. Χρειάζεται ένα συντονισμένο πρόγραμμα που θα δίνει κίνητρα για τις επενδύσεις στις επιχειρήσεις με την ε, έρευνα και την δημιουργία δράσεων που θα λαμβάνει υπόψη την, πρόσθετη, την παραγωγή πρόσθετης αξίας Ιδιαίτερα τα 115 ε, ε, δις ε, ευρώ πρέπει μέσα σε αυτό το πλαίσιο να θεωρηθούν ανεπαρκή. Τι γίνεται σε σχέση με τα υφιστάμενα σχέδια. Για τις επενδύσεις αυτές είναι συμπληρωματικές ή εντάσσονται στα προγράμματα του ορίζοντα 2020 κτλ. Απ' την άλλη πλευρά είχε προαναγγείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτά είναι αυτά τα οποία θα αναγγελθούν. Παρακαλώ να προσέξετε σε σχέση με την ε, παρέμβασή σας ολοκληρώθηκε ο χρόνος ή στη συνέχεια. Ο κύριος Λούκε από την ECR. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριοι επίτροποι, Μία ερώτηση προς τον κύριο Ντομπρόσκης ε, για τα 315 δις ε, πακέτο επενδύσεων. Μόχλευση θέλετε να πετύχετε 1 προς 15, 15 πλάσια. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος των επενδύσεων θα πρέπει να το υπομισθούν οι ιδιώτες επενδυτές. Αυτό θα το κάνουν όμως οι ιδιώτες επενδυτές μόνο όταν θα έχουν τη δυνατότητα αποκόμισης κερδών από αυτές τις επενδύσεις. Συνολικά δηλαδή ώστε να μπορούν να χρηματοδοτηθούν, να ε, αποσβεστούν αυτές οι επενδύσεις. Σε σχέση με την κατάσταση κρίσης αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά το ότι οι πολίτες στα κράτη κρίσεων θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι την προσέγγιση προσπάθεια αυτή. Δηλαδή για την ε, εκμετάλλευση και την χρήση των υποδομών για παράδειγμα. Ώστε επιπρόσθετα θα επιβαρυνθούν αυτοί οι πολίτες σε κράτη κρίσης τα επόμενα χρόνια. Αυτό το οποίο πουλάει ως δώρο προς τους πολίτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια επιβάρυνση φορολογική για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί αυτή η επένδυση. Δεύτερη ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει σαν μέσα από αυτά τα κίνητρα να δημιουργούσε πρόσθετες επενδύσεις. Αυτό όμως δεν διασφαλίζεται με κανένα τρόπο. Δίνει κίνητρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα υπάρξει πιθανότητα μια μετακύληση και μια μετάθεση προγραμμάτων και σχεδίων επενδύσεων που θα βρίσκονται στο όριο της κερδοφορίας ή της μη κερδοφορίας. Και έτσι σε σχέση με τις βέβαιες σίγουρες επενδύσεις ε, θα υπάρχει διαφοροποίηση. Δεν θα είναι λοιπόν 315 αυτά τα δισεκατομμύρια που θα χρησιμοποιηθούν ενιαία προς αυτό το στόχο. Κυρία Χάρκιν παρακαλώ στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Η πρώτη μου ερώτηση λέει η κυρία Χάρκιν έχει να κάνει με την ε, φτώχεια. Γίνεται λόγος για τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού που αυξάνεται από 8,7 εκατομμύρια πολίτες και συνεχίζει να αναπτύσσεται αυτός ο αριθμός ε, των ατόμων αυτών. Στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε ότι περισσότεροι κοινωνικοί δείκτες πρέπει να χρησιμοποιούνται και επίσης γίνεται λόγος για την εισαγωγή αυτών των δικτών στη χρήση και την εφαρμογή. Πρώτη ερώτηση, μπορείτε να είσαστε πιο συγκεκριμένοι για αυτούς τους κοινωνικούς δείκτες και δεύτερον, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι κοινωνικοί κοινωνικοί δείκτες σε αυτές τις διεργασίες για να αντιμετωπιστεί το θέμα της φτώχειας και της ε, μισθολογικής φτώχειας ώστε να αντιμετωπιστούν οι σοβαρότατες ε, ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών. Η δεύτερη ερώτησή μου και αυτή αφορά τις ανισορροπές ε, σχέσεις, τις ανισορροπίες που υπάρχουν. Γίνεται λόγο στην έκθεση ότι κάποια κράτη-μέλη ότι δηλαδή τα πλεονάσματα σε κάποια κράτη-μέλη δεν μειώθηκαν επαρκώς σε σχέση με την μεγάλη προσπάθεια αντιστάθμισης των οικονομικών ανισορροπιών. Επίσης λέτε ότι τα πλεονάσματα δεν θέτουν ε, τις ίδιες προκλήσεις ε, όσον αφορά την βιώσιμη κατάσταση χρέους ε, για τα κρατημέλη. Τι κάνετε λοιπόν για να αντιμετωπίσετε την πρόκληση των πλεονασμάτων στους λογαριασμούς και μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς μπορούν να συνεισφέρουν οι δράσεις αυτές στην επίτευξη του στόχου. Ευχαριστώ κυρία Τάισεν, ελπίζω ότι θα μπορέσετε σε τρία λεπτά να απαντήσετε αυτές τις ερωτήσεις. Um, Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, προς τον κύριο Σάντ, σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είμαι ικανοποιημένη που και στο Κοινοβούλιο τρέβεται μεγάλη προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί στην τελική ανάλυση το ξέρουμε εδώ και χρόνια είναι η κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης και κατά το παρελθόν 85% των νέων θέσεων απασχόλησης δημιουργούνται στους κόλπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτό το ποσοστό έχει μειωθεί πλέον. Αυτό τι σημαίνει ότι αναλογικά επιβαρύνονται πιο πολύ και δυσκολεύονται πιο πολύ. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε για να επιλύσουμε τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να έχουν ανάγκη θέσεις υπαλλήλου ε, ε, και να τους προσλαμβάνουν και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα σε σχέση με τους μεγάλους ομίλους. Είναι μεγαλύτερη η δυσκολία τους να έχουν πρόσβαση σε δάνεια, σε πιστώσεις, σε ρευστότητα σε σχέση με την πρόσβαση λοιπόν στην κεφαλαιοχική αγορά. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το, δώσουμε, το επιλύσουμε ως πρόβλημα στα πλαίσια και του προγράμματος Small First. Μία άλλη ερώτηση τώρα προς την ίδια κατεύθυνση. Η αντίστροφη φτώχεια, η κοινωνικός αποκλεισμός, οι κοινωνικοί δείκτες. Δεν έχω πολύ χρόνο να απαντήσω. Πώς θα τους χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τους δείκτες αυτούς. Ακριβώς αυτό πρέπει να βρούμε. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν όχι μόνο επειδή θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει σε κάθε χώρα, αλλά επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι αν ε, κινηθούν προς λάθος κατεύθυνση οι κάποιοι κοινωνικοί δείκτες, όπως για παράδειγμα η ενεργία, η ενεργία των νέων, υπάρχει ανισορροπία. Και η ανισορροπία αυτή θα πρέπει να καταπολεμηθεί και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα οικονομικής διακυβέρνησης. Δεν ξέρουμε όμως ακριβώς πώς θα χρησιμοποιηθούν. Σημαντικό θα είναι να αναπτυχθούν κατόφλια και προ την κατεύθυνση λοιπόν αυτή θα κινηθούμε του επόμενου μήνε. Σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να τεθούν τα κατόφλια. Γιατί τα κατόφλια, ε, οι δείκτε αυτοί θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και κατά χώρα, αναχώρα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ιδιαιτερότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε τις επόμενες εβδόμες και ασφαλώς και θα διαβουλευτούμε στην διαδικασία αυτή και με το Κοινοβούλιο αλλά και με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο. Πολλά μπορεί να μπει κανεί σε 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Θα δώσω το λόγο στον, στον, Επίτροπο για την αύξηση των πλονασμάτων στην Ευρώπη σε σχέση με το 2008-2014. Προφανώς αποτυπώνει το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη πιστωτές από πλευράς τους δεν έχει μειωθεί αρκετά το πλεόνασμα σε ό,τι αφορά τις οικονομίες που είναι χρεωμένες. Τι αποτυπώνει λοιπόν αυτό. Οικονομικές ε, ε μη αναποτελεσματικότητες σε ό,τι αφορά τη ζήτηση και την προσφορά σε ό,τι αφορά τα αρνητικά μετακύληση, την αρνητική μετακύληση προς τους εταίρους. Αυτή λοιπόν το θέμα θέλει να καταπολεμήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αποτελεσματικές επενδύσεις για να υποστηρίξει την εγχώρια ζήτηση και την ανάπτυξη και προφανώς αυτό αποτελεί βασική προτεραιότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στις χώρες πιστωτές. Και αυτό είναι το μήνυμα που αναπτύσσουμε από κοινού με τον κύριο Ντομπρόφσκη για το σχέδιο προπολογισμού. Ευχαριστώ κύριε Ντομπρόφσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε επικεντρωθώ στις ερωτήσεις που αφορούν ε, το πακέτο των επενδύσεων, που ήταν αρκετές. Πρώτα, η ερώτηση της κυρίας ε, Ριμπέρο για το κατά πόσον αυτά τα 300 δις ε, επαρκούν. Να σας δώσω μια εικόνα πώς προέκυψε το ποσό του πακέτου. Αν δούμε τις βιώσιμες επενδύσεις, οι οποίες ε, έγιναν και πολλά χρόνια πριν από την κρίση, είδαμε ότι είχαμε ε, επενδύσεις στις τάξεις του 20-21% του ΑΕΠ ε, στην Ευρώπη πριν από την κρίση ανεβήκαμε στα χρόνια της ε, ανάκαμψης ε, και αυτό φυσικά αντανακλούσε και κάποιες ε, αγορές στεγαστικών και κατασκευών σε κάποιες χώρες μέλη που ήταν ιδιαίτερα αυξημένες και έκτοτε έχουν πέσει ουσιαστικά οι επενδύσεις. Είναι πολύ σημαντική η μείωση και είμαστε και πάλι στο 20 με 21% του ΑΕΠ. Και η έλλειψη αυτή είναι κάπου μεταξύ 230 και 370 δις ευρώ και γι' αυτό ακριβώς ανακοινώθηκαν 300 ε, δις ευρώ ή 315 και αυτό περίπου βρίσκεται ε, μεταξύ αυτού του φάσματος των 230 και των 370. Να σας πω δηλαδή πώς προήλθαν αυτά τα 300 δις. Τώρα, για την ερώτηση του κυρίου Λούκε, για το κατά πόσον αυτό το πακέτο επενδύσεων θα καταλήξει τελικά να είναι ε, κάποιος ε, ε, κρυφός φόρος που θα επιβάλλουμε στους πολίτες. Αναφερθήκατε στο ποσοστό της μόχλευσης που σημαίνει σαφέστατα ότι η ιδέα αυτού του πακέτου περιορίζει το ποσό των δημοσίων κονδυλίων προκειμένου να έχουμε περισσότερες επενδύσεις από ιδιωτικά κονδύλια. Και αυτό είναι το σκεπτικό. Άλλωστε, με τη βοήθεια των ιδιωτικών κονδυλίων θα μπορέσουμε να έχουμε και τη δυνατότητα για ε, απορρόφηση ε, πρώτου βαθμού. Τώρα, για να απαντήσω και στο πρώτο τμήμα της ερώτησής σας, η μία από τις επικρίσεις που απευθύνονται τώρα προς την Ευρώπη και στα κράτη-μέλη είναι ότι έχουμε πάρα πολύ χαμηλά επιτόκια, επιτόκια ρεκόρ στις περισσότερες χώρες και παρόλα αυτά δεν εκμεταλλευόμαστε αυτή την ευκαιρία για να επενδύσουμε. Είναι σαφές ότι οι επενδύσεις θα έχουν κάποιο κόστος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε ε, άμεσα μέσω του προϋπολογισμού, είτε μέσως, αλλά τελικά κάποιο θα πληρώσει για τι επενδύσει, αν απλώ και μόνο είναι ιδιωτικές επενδύσεις. Το ερώτημα όμω είναι αν τα ωφέλη αυτή τη επένδυση αν έχουμε για παράδειγμα μια αποδοτική ενεργειακή κοινότητα, αν έχουμε ενεργειακή απόδοση ή αν έχουμε επενδύσεις κάπου αλλού. Εάν ε, τα ωφέλη των επενδύσεων είναι μεγαλύτερα από το κόστος της επένδυσης και αυτό είναι και το όλο σκεπτικό των επενδύσεων εν γέννη. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν να επιλέξουμε και τα κατάλληλα προγράμματα προς επενδύσεις που θα μας οδηγήσουν σε ωφέλη και φυσικά να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη και τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση αυτού του πακέτου, να μην είναι απλώς ε, μια πολιτική διαμεσολάβηση, αλλά να είναι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται ε, με κατάλληλο τρόπο, να διατεθούν και κονδύλια σε μικρές επιχειρήσεις και είναι σαφές ότι σίγουρα αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε και θα πρέπει τα ωφέλη ε, της επένδυσή μας να αποδώσει. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει το κόστος. Δεν απαντάτε κύριε Ντομπρόσκη, ο κύριος ναι. Λούκε. Πολύ σύντομη απάντησή σας παρακαλώ. Όπως σας είπα, βεβαίως και εξαρτάται από το πρόγραμμα, αλλά τελικώς το κόστος με τον ένα με τον άλλο τρόπο κάπως θα πληρωθεί. Θα είναι δημόσια ε, κονδύλια μέσω των φορολογουμένων είτε μέσω των ιδιωτικών επιχειρήσεων που θα επενδύσουν και θα πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο της επένδυσής τους. Αυτό που έχει σημασία είναι τα ωφέλη της επένδυσης να είναι μεγαλύτερα από το κόστος. Αυτό είναι το όλο σκεπτικό της επένδυσης. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στον τρίτο γύρο. 1,5 ε, λεπτό για τους κοιόδης εισηγητές και 10 λεπτά ε, συνολικά για τους επιτρόπους για να απαντήσουν σε ερωτήσεις σας. Σας παρακαλώ μην ε, αγορεύετε ε, στις ερωτήσεις που θα θέσετε. Ο κύριος Τόιρερ από τους Φιλελευθέρους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμη επίτροπη. Μία ερώτηση προς εμάς κύριε Ντομπρόφσκης. Στην Λετωνία πραγματικά εντυπωσιακό εξηγιαντικό πρόγραμμα ακολουθήσατε. Άλλες χώρες αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όμως. Πιστεύετε ότι η Γαλλία και η Ιταλία θα πρέπει να πάρουν το πεπρωμένο στα χέρια τους και με παρόμοιες μορφές όπως η Λετωνία να δράσουν. Δεν είναι θέμα δικαιοσύνης. Οι μικρές χώρες που υλοποίησαν τις ε, υποχρεώσεις τους, άλλες όμως ε, να δυσκολεύονται, δεν είναι ε, ανισό αυτό. Και στο θέμα της ανταγωνιστικότητας και των μη ισόρροπων σχέσεων ε, πλεονάσματα εξαγωγικά ε, υφίστανται επικρίσεις. Όμως ε, εξαγωγικά πλεονάσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά δεν απαιτούνται αν θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα σύμφωνο ανάπτυξης και στη Γερμανία κάθε γερμανικό αυτοκίνητο που εξάγεται 40% της δημιουργίας ε, πρόσθετης αξίας προέρχεται από όμορα κράτη. Δηλαδή μια τέτοια εξαγωγή είναι θετική όχι μόνο για τη Γερμανία αλλά για το σύνολο της Ευρώπης. Πώς κάτι τέτοιο θέλετε να το πετύχετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεδομένων των διαφορετικών απόψεων των διαφορών που είναι ευδιάκριτες πλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Madam starting. Τάισεν, εσείς, παρακαλώ. Okay, we'll continue with the questions. Να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις, προκειμένου να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται. Η κυρία Μακιντάιρα από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω πόσο ισχυρή είναι η δέσμευση στην ε, ε, μελέτη ετήσιας ανάπτυξη προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη θέσεων απασχόληση. και χαίρομαι ιδιαίτερω που υπάρχει νέα δέσμευση για τι διαθετικέ μεταρρυθμίσει. Η Επιτροπή Στάισεν μας είπε με σαφήνεια ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσει και ότι θα πρέπει να περάσουν οι μεταρρυθμίσεις αυτές για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον μια μελέτη της, της, της ε, Παγκόσμιας Τράπεζας σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις το 2015 και για την ε, αποτελεσματικότητά τους. Αξιολογήθηκε λοιπόν το κανονιστικό πλαίσιο για όλες τις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η χώρα μου, είναι η δεύτερη διαπίστωση μεγάλη μου χαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατάταξη. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό τα κρατημέλη να διδάσκονται τα μένα από τα δέν, προκειμένου να υπάρχει συνολικά ανταγωνιστικό κλίμα σε παγκόσμιο προσκήνιο. Προκειμένου να επαναφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις θέσεις απασχόλησης. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, μπορείτε να μας δώσετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για το πού θα χρειαστεί να κάνουμε μεταρρυθμίσεις και πώς θα το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ. Μιγκουέλ Μιβιέγκας από την ΚΟΕ. Ε, Αυτή η ανάλυση, ετήσια ανάλυση της ανάπτυξης, θεωρούμε εμείς, δεν δίνει τίποτα το καινούριο. Είναι συνέχεια της παλαιάς πολιτικής. Περικοπές του κοινωνικού κράτους, απελευθέρωση των αγορών αναμονή και πίστη ότι η αγορά θα λύσει όλα τα προβλήματα. Και όπως είναι προβλέψιμο όλα θα παραμείνουν στην ίδια κατάσταση για να μην πούμε στη στασιμότητα που θα συνεχίσουν οι νέοι να είναι άνεργοι και χωρίς μέλλον. Για τις επενδύσεις θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια. Πρώτο, θα ήθελα να μου πείτε Πώς διαφοροποιούνται αυτές οι επενδύσεις σε σχέση με το σύμφωνο σταθερότητας που ξεκίνησε το 2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τότε ήταν 120 δις ε, ευρώ και βασιζόταν στο ίδιο παραμύθι της, ε, του πολλαπλασιασμού των ευεργεσιών. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η αξιολόγηση αυτού του Συμφώνου σταθερότητας που ξεκίνησε το 2012 από πλευρά σα. Από την άλλη πλευρά σε σχέση με την κλίμακα. Θα ήθελα επίση ε, να πω ότι είναι απόλυτα ανεπαρκής. 20% μείωση έχουμε κατακρίνηση των επενδύσεων ε, και σε σχέση με τις, ε, την, ε, τις προσδοκίες μέσα σε, στο χρονικό πλαίσιο είναι ανεπαρκέστατο. Και τέλος, όσον αφορά μια ερώτηση για τη δυνατότητα των κρατών να μπορέσουν να ενταχθούν και να χρησιμοποιήσουν αυτό το ταμείο, αυτή τη δυνατότητα. Πώς εξηγείται ότι οι δαπάνες οι εθνικές πάνε, υπολογίζονται στο έλλειμμα και πώς υπάρχει τη δυνατότητα τα κονδύλια, τα ταμεία. Πρέπει να σας διακόψω δυστυχώς, έληξε ο χρόνος σας. Και τώρα ο Νεοκλής Ηλικιώτης παρακαλώ, από την Ενωτική Αριστερά, έχετε τον λόγο. Η Επισκόπηση Ανάπτυξης μιλά για περαιτέρω λιτότητα, για θεσμοθέτηση της δημοσιονομική πειθαρχίας και επενδύσεις που μπορούν να απέχουν από τη στήριξη ανάκαψης τη πραγματική οικονομία. Την ίδια ώρα, όπω αναφέρθηκε, οι αριθμοί των μακροχρόνων ανέργων βοού το πρόβλημα της νεανικής ανεργίας μετατρέπεται σε ένα από τα μεγαλύτερα της Ένωσης. Ο νότος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποβιομηχανοποιείται. Οι μισθοί καρταρέου, τα δικαιώματα των εργαζομένων δέχονται ανηλαιή επίθεση. Οι εργασιακέ σχέσει απορριθμίζονται, παραβιάζονται ακόμα και θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι πολιτικέ λιτότητε και η ανεξέλεκτη απορρίθμιση τη αγορά επιβάλλονται μέσω τη Τρόικα στι χώρε του Νότου και δυστυχώ η ετήσια ε, ε, επισκόπηση ανάπτυξη επιμένει η Επιτροπή στις ίδιες συνταγές χωρίς να αντιλαμβάνεται το παράδοξο του να προτείνονται οι αιτίε των προβλημάτων ω οι λύσει τους. Ερωτώ τον κύριο Αντιπρόεδρο, πώ μπορείτε να διασφαλίσετε τον κοινωνικό διάλογο που τόσο πολύ διακρίσετε στα κράτη-μέλη με μνημόνιο τη στιγμή που η Τρόικα πιέζει τις κυβερνήσεις για, για βίαιη μείωση του εργατικού κόστου και για λιτότητα η οποία συντείνει ακριβώς την απορρίθμιση των εργασιακών θεσμίων. Ερωτώ την κυρία Επίτροπο Τάισεν, στην ακρόαση σα, κατά τη διάρκεια ε, τη ακρόαση στο Κοινοβούλιο, τονίσετε ότι χρειάζονται να ενταχθούν κοινωνικοί δείχτε. Σήμερα είπατε πάλι για κοινωνικού δείχτε, που, μερικοί από αυτού εντάχθηκαν ε, στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όμω, η κατάσταση στον Νότο και στις χώρες του μνημονίου είναι σημαντική. Θέλουμε, κυρία Τάισεν, κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις ό,τι αφορά την ένταξη των κοινωνικών δίκτων. Ε. Συγγνώμη, πρέπει να σας διακόψω. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μουσκοβισή. Δεν θέλετε το λόγο. Θα Ξεκινήσουμε με την κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η κυρία Μάκιντάιερ μου έκανε ερώτηση και ο τελευταίος ε, συνάδελφος από την Ελλάδα. Τι μεταρρυθμίσεις λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε, ρωτάτε κυρία Μάκιντάιερ. Νομίζω ότι έχουμε ένα ολόκληρο πλωστάσιο. Έχουμε τους στόχους του 2020, Ευρώπη του 2020 με πέντε μεγάλους ε, τους στόχους, προτεραιότητες και τις ε, εμβληματικές ε, πρωτοβουλίες. Έχουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση σύντομα. Θα μπορέσει και το Κοινοβούλιο λοιπόν να αποφαθεί και σίγουρα θα χρειαστούμε τις προτεραιότητες αυτές. Έχουμε τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισοτήτων όταν έχουμε την αίσθηση ότι στις ε, κάποιες χώρες υπάρχουν σημαντικά προβλήματα, μπορούμε να κάνουμε την εισβάθος ανάλυση και στη συνέχεια είτε να περάσουμε στην ε, συγκεκριμένη διαδικασία ή να κάνουμε συστάσεις ανά χώρα σε ό,τι αφορά το εγχείρημα της Ευρώπης 2020 και στην τελική ανάλυση το θέμα είναι τα κρατή-μέλη γιατί πιο πολλές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν στα κράτη-μέλη και έχουν αρμοδιότητα για αυτές τα κράτη-μέλη. Άρα προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε τα κράτη-μέλη προκειμένου να τους δείξουμε ποιες διαφορές υπάρχουν και που μπορούν να πάνε καλύτερα. Και χρειάζεται και το πακέτο επενδύσεων και θα πρέπει να κοιτάξετε στην τρίτη, στον τρίτο πυλώνα όπου αναφέρεται οι μεταρρυθμίσεις. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα προσκόμματα για τις επενδύσεις. Δεν έχουμε μόνο το πακέτο 300 350 δισεκατομμυρίων, έχουμε και τον τελευταίο πυλώνα μέσα στο πακέτο που αφορά τις διαστατικές μεταρρυθμίσεις. Έχουμε και την ατζέντα για την ιστορική αγορά που θα πρέπει να ολοκληρωθεί και το συνολικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής περιλαμβάνει μια ατζέντα για τις θέσεις απασχόλησης, την ανάπτυξη και την ε, κοινωνική ισότητα και νομίζω ότι όλη αυτή την ατζέντα πρέπει να εξετάσουμε και να βγάλουμε όποια εργαλεία μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν οι απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να βελτιωθεί η, τη θέση απασχόλησης σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς δείκτες. Το ερώτημα του κ. Σιλικιώτη. Νομίζω ότι απάντησα σε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Οι κοινωνικοί δείκτες έχουν συμπεριληφθεί και σε όλη την ανάλυση δίδεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για την κοινωνική κατάσταση στα κράτη-μέλη και στο μέλλον το έχουμε συμφωνήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσουμε και θα συμπεριλάβουμε τους κοινωνικούς δείκτες ως ισότιμους δείκτες. Θα καθορίσουμε κατόφλια και η άσκηση αυτή θα ξεκινήσει σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ντομπρόφσκης. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα επικεντρωθώ στα ερωτήματα του κυρίου Τόιερ σε ό,τι αφορά τη Γαλλία και την Ιταλία και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα πλεονάσματα των ισολογισμών. Όπως αναφέρθηκα και στα εισαγωγικά μου σχόλια, έχουμε 7 χώρες καταρχάς όπου στον τρέχοντα κύκλο οικονομικής διακυβέρνησης θεωρούμε ότι υπάρχει κίνδυνος αστάθειας και σε ό,τι αφορά το σύμφωνο σταθερότητας. Έχουμε τρεις χώρες που είναι σε μεγάλο κίνδυνο, η Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο. Η Γαλλία σε ό,τι αφορά την πρόοδο για τη συμμόρφωση με τις συστάσεις του Συμβουλίου για τη διαδικασία υπερβολικών πλεονασμάτων, Ιταλία και το Βέλγιο σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις με το δημόσιο χρέος και θέματα βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Αλλά, όπω ανέφερα, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε επιστολές και από τις τρεις χώρες αυτές, όπου εκφράζονται η δέσμευσή τους για τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις και η προθυμία τους να κάνουν δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε πιο πολύ χρόνο στις χώρες αυτές μέχρι την Άνοιξη προκειμένου να μπορεί μέχρι την Άνοιξη να αξιολογήσει την κατάσταση για τα, τρία χρο... για τα τρεις χώρες αυτές βάσει συγκεκριμένων δεδομένων και στοιχείων. Και λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανέλθει στο θέμα αυτό την Άνοιξη. Με όλες τις δυνατότητες σε ό,τι αφορά την πολιτική, αλλά και με πιο ακριβή αριθμητικά στοιχεία, με ανάλυση ελπίζουμε μακροοικονομική από, ε, από την εισβάθο ανάλυση χώρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πλεονάσματα των ισολογισμών. Αναφερθήκατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τρέχον ε, πλεόνασμα, το οποίο ασφαλώς είναι καλό. Η Γερμανία, η Γερμανία θεωρώ, κατά πάσα πιθανότητα είναι η χώρα που συνεισφέρει πιο πολύ από όλες στο πλεόνασμα. Ωστόσο, για τις μακροοικονομικές διαδικασίες διακυβέρνησης στο σχετικό μηχανισμό έχουμε θέσει μακροοικονομικούς δείκτες και κατόφλια, κατώτατες τιμές. Και τώρα σε ό,τι αφορά τα πλεονάσματα είναι 6% του ΑΕΠ για τρία χρόνια κατά μέσο όρο και αν μια χώρα υπερβεί το ποσοστό αυτό μπορούμε να αποφασίσουμε να εξετάσουμε σε βάθος το θέμα αυτό. Να κάνει λοιπόν εις βάθος ανάλυση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη Γερμανία για τα πλεονάσματα. Και αυτό ενδεχομένω να έχει δύο συνέπειες. Το θετικό στοιχείο είναι η μεγάλη ανταγωνιστικότητα της χώρας, το αρνητικό είναι η ασθενή εγχώρια ζήτηση και επένδυση. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διεξαγάγει εις βάθος ανάλυση και θα σας παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μουσκοβισή. Ναι. Θα ήθελα καταρχάς να καθησυχάσω τον κύριο Τόιρερ. Δεν ξέρω, μήπως δεν κατάλαβα καλά. Αλλά δεν υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις που έχουμε λάβει ε, με τον κύριο ε, Βοντρόφσκης, όπως ακούστηκε, ελήφθησαν σε πλήρη αρμονία, χωρίς κανένα δισταγμό, διότι πιστεύουμε και η μεν και η δε ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τους κανόνες, κάτι που θα κάνουμε και ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση των διαφόρων χωρών που το κάναμε και να συνεχίσουμε να πιέζουμε, κάτι το οποίο θα κάνουμε και δεν θα χαλαρώσουμε ε, έτσι ελαφρά την καρδία. Ε, υπάρχει ένα σύμφωνο το οποίο λαμβάνουμε φυσικά υπόψη, λαμβάνουμε υπόψη και τις προσπάθειες φυσικά που κάνει ο καθής και να σας υπενθυμίσω ότι και για την Ιταλία και για το Βέλγιο και για τη Γαλλία οι τρεις ε, ε, πρωθυπουργοί απέστειλαν επιστολές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να λαμβάνουν δεσμεύσεις και περιλαμβάνει και χρονοδιάγραμμα. Χρονοδιάγραμμα στο Συμβούλιο Υπουργών, ψηφοφορίας ε, και ούτω καθεξής και ε, χρονοδιάγραμμα παρουσίασης των συνεπειών της τάδε μεταρρύθμισης επί του προγράμματο. Μην νομίζετε λοιπόν ότι είναι τσιγαρόχαρτο αυτό το οποίο περνάνε οι επίτροποι μεταξύ τους και δεν έχουν συμφωνήσει επί τίποτα. Είναι πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τώρα, στον κύριο Βιέγκας για να συγκρίνουμε το τι έγινε το 2012 και το τι αποφασίστηκε τώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ένας πλήρης απολογισμός των όσων ε, συμφωνήθηκαν το 2012. Ναι, δεν ήταν μεν η πλήρης επιτυχία, αλλά δεν ήταν και η πλήρης αποτυχία που παρουσιάζουν κάποιοι. Ε, αν για παράδειγμα ε, σταθώ στο παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ε, αυξήθηκε κατά 5% το κεφάλαιο της τράπεζας και αυτό ισχύει γενικότερα και για τις επενδύσεις. Αλλά βέβαια κάποιοι μηχανισμοί δεν λειτουργήσαν όσο θα έπρεπε, ε, παραδείγματος χάρη τα ομόλογα έργου, τα οποία έμειναν σε πειραματικό στάδιο και τα οποία εξορισμού δεν ήταν αυτό το οποίο θέλαμε, θέλαμε να περάσουμε στο επιχειρησιακό στάδιο και η διαφορά τώρα είναι όσον αφορά την ταχύτητα των αποφάσεων και την ταχύτητα εφαρμογής που είναι αποφασιστική σημασία 300 ε, ε, δις σε τρία χρόνια είναι πάνω από 120 σε 1,5 χρόνο φυσικά και όλα αυτά ε, θα πρέπει να γίνουν και με συγκεκριμένους στόχους, διότι θέλουμε να ευνοήσουμε επενδύσεις οι οποίες θα μας δημιουργήσουν ανάπτυξη στο μέλλον και θα μας επιτρέψουν να έχουμε, για παράδειγμα, ε, ψηφιακή ανάπτυξη, ενέργεια, μεταφορές, οτιδήποτε άλλο, ε, ε, οτιδήποτε είναι η οικονομία της γνώσης και όλα αυτά θεωρούμε ότι θα έχουν πολύ πιο σημαντικές συνέπειες στην ανάπτυξη και λόγω της βαρύτητά τους αλλά και για τη ταχύτητα εφαρμογής. Ευχαριστώ. Να περάσουμε τώρα στον τέταρτο γύρο, ερωτήσεις ενός λεπτού και εννέα λεπτά για τους επιτρόπους για να προσπαθήσουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μωρίς Σαρτιέ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακούσαμε πολλά για σταθερότητα και για δυναμική. Θα ήθελα να θέσω τις εξή ερωτήσεις στους Επιτρόπους. Πρώτη ερώτηση. Έχετε συμπεριλάβει στις προβλέψεις σας και την εξέλιξη της απασχόλησης, διότι γνωρίζουμε ότι από τώρα μέχρι το 2020 15% ε, των θέσεων εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης θα εξαφανιστούν και θα χρειαστούμε 15% θέσεων εργασίας υψηλού επίπεδου εξειδίκευσης. Ε, Έχετε ακολουθήσει ε, λογική σταθερής γεωμετρίας ή μεταβλητής γεωμετρίας. Δεύτερη ερώτηση. Οι γυναίκες οι οποίες έχασαν τη θέση εργασίας τους ε, στη διάρκεια της κρίσης, τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε προκειμένου να βρείτε αυτούς τους εργαζομένους που έχασαν τις θέσεις εργασίας τους και πλήγησαν ιδιαίτερα κυρίως οι γυναίκες λόγω ε, του χαμηλού μισθού και των επισφαλών συμβάσεων εργασίας. Τρίτη ερώτηση, οι νέοι και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έχετε προβλέψει να υπάρξει κάποια παρακολούθηση προκειμένου να μετρήσετε τις ε, συνέπειες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ε, ως προς την επιστροφή των νέων στην αγορά εργασίας και μάλιστα μια βιώσιμη επιστροφή. Ευχαριστώ από τους Πρασίνους, ο κύριος ε, Γκουστασόν. Ευχαριστώ. Έχω την εντύπωση ότι παρουσιάστηκε αυτή η έκθεση χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη να οι αρνητικότατες προοπτικές υπό τις οποίες ζούμε στην Ευρώπη τώρα προτείνουν να συνεχιστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ υπάρχει αρνητική επίπτωση για την ανάκαμψη και για το πακέτο δέσμης μέτρων για τις επενδύσεις υπάρχουν σημαντικές αμφιβολίες αν θα λειτουργήσουν όλα σωστά ή όχι. Έχω δύο ερωτήσεις για τα θέματα που θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Δηλαδή την μείωση της, ε, του και τις μήνες. Κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη αρνητική επίπτωση όσον αφορά την ε, ζήτηση και όσον αφορά την ανάκαμψη και ο ΣΑ το ανέφερε σε μια έκθεση αυτό το Σεπτέμβριο ήδη από πλευρά του. Πρώτη ερώτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάποια αξιολόγηση για τις αρνητικές επιπτώσεις ε, όσον αφορά την ανάπτυξη κάποιων των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας και των αρνητικών ε, επιπτώσεών τους. Για τον Επίτροπο Μοσκοβισή, στην ακρόασή σας υπό, τότε που είσαστε υποψήφιος ε, ε, επίτροπος είχατε πει ε, διάφορα πράγματα. Ερώτηση, το σενάριο αυτό το οποίο είχατε παρουσιάσει, πότε θα θεωρείτε ότι πραγματικά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η σοβαρή αρνητική οικονομική εξέλιξη και σε σχέση με το πώς θα χρησιμοποιηθεί η ελαστικότητα, θα ήθελα όμως να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες πώς οι ανισορροπίες υπολογίζονται, διότι αυτό δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και πρέπει να μας το πείτε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροντρίγκε παρακαλώ. Καλημέρα σας. Θεωρώ ότι η επισκόψη για την ετήσια ανάπτυξη βελτίωσε την προσέγγιση όσον αφορά την προσφορά. Αναγνωρίζετε ότι η παράμετρος της προσφοράς δεν είναι μόνο το θέμα των μεταρρυθμίσεων, είναι επίσης και ζήτημα επενδύσεων που χρειάζονται, κυρίως επενδύσεων είναι μια πρόοδος αυτή, παρότι πιστεύω ότι πάρα πολλά πρέπει να συζητηθούν ακόμα για το πώς οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν αλληλεπίδραση με τις μεταρρυθμίσεις ώστε να υπάρξει δυνατότητα να προαχθεί ανάπτυξη. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό, ε, ε, μια σημαντική έλλειψη και αυτό είναι σε σχέση με τη ζήτηση. Νομίζω αγνοεί ή υποβαθμίζει την ε, ε, απουσία ζήτησης που υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως πίσω από αυτή την κατάσταση έλλειψη ζήτησης στην Ευρώπη έχουμε ανισότητες που αυξάνονται μέσα στα ίδια τα κράτη-μέλη μας και μεταξύ όμως και των κρατών μελών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στραγγαλίζει τη ζήτηση στην Ευρώπη. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τα αίτια, οι ρίζες του προβλήματος. Και τα αίτια, οι ρίζες του προβλήματος συσχετίζονται με το την μισθολογική πολιτική, τη φορολογική πολιτική, αλλά επίσης και πολύ διαφορετικούς όρους υπό τους οποίους γίνονται επενδύσεις. Το πρόγραμμα επενδύσεων είναι δεδομένο, όμως το πρόγραμμα επενδύσεων πρέπει να σχεδιαστεί ώστε αυτές οι διαφορετικές προϋποθέσεις και όροι για επενδύσεις σε σχέση με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μία ερώτηση προς την Επίτροπο ε, Τάισεν. Κάνατε λόγο για κοινωνικό διάλογο, λέει η κυρία Βάνα. Πιστεύετε ότι οι κοινωνικοί εταίροι και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει ενδυναμωμένα να εμπλακούν στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, ιδιαίτερα και η κοινωνία των πολιτών, όπως κατά το παρελθόν, κατά την προηγούμενη περίοδο, είχε προαναγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στο Στρασβούργο είχαμε και ένα ψήφισμα το οποίο εγκρίναμε την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά. Οι πολίτε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγα, δεν πρέπει να μας βλέπουν μόνο ως εκείνους που επιβάλλουν νεοφιλελεύθερες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις, αλλά που τους δίνουμε τη δυνατότητα συνδιαμόρφωσης ε, των πραγμάτων. Διότι αυτές οι ε, μεταρρυθμίσεις έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις και είχαν αρνητικές επιπτώσεις στους πολίτες. Ελαστικοποίηση των ωραρίων ε, και όρων απασχόλησης, περικοπές μισθολογικές, επιπτώσεις που ήταν αποτελέσματα των πολιτικών της Τρόικας. Πώς θα διασφαλίσετε, ερώτησή μου, αυτές οι προαναγγελθήσεις ε, ε, κατευθυντήριες γραμμές να οδηγήσουν στη συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών. Και ποια κονδύλια και μέσα θα διαθέσετε για να επιτευχθεί αυτό. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Τάισεν για να απαντήσει παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε, να προσπαθήσω να απαντήσω εν συντομία, όπως μου ζητήσατε. Το πρόβλημα που αναφέρατε κυρία Μωράν Σματιέ είναι σημαντικό γιατί ξέρουμε ότι όσοι δεν έχουν καλή εκπαίδευση είναι αυτοί που βγαίνουν από την αγορά εργασία ε, πρώτοι και δεν μπορούν να ξαναμπούν εύκολα. Θα πρέπει λοιπόν και οι νέοι αλλά και οι πρεσβύτεροι να φροντίσουμε να έχουν καλή εκπαίδευση, καλά προσόντα και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και πρωτοβουλία για την ε, καταπολέμηση της ενεργείας των νέων εδώ λοιπόν εστιαζόμαστε πραγματικά στην προσόντα, στην επαγγελματική κατάρταση. Πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και στο πακέτο επενδύσεων όπου μιλάμε για εκπαίδευση. Διευκρινίζουμε ότι πρόκειται και για vocational training, επαγγελματική κατάρτιση. Πραγματικά μεγάλη σημασία δεν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σκέλος αυτό. Σε ό,τι αφορά τα, ποια είναι η συνέχεια και η παρακολούθηση για το κατά πόσο ξέρουμε αν υπάρχουν αποτελέσματα των δράσεών μας. Χθες στο Παρίσι παρέστησα σε μια εκδήλωση για ένα λειτουργικό πρόγραμμα για το Ταμείο στη Γαλλία όπου και τόνισα ότι δεν υπάρχουν μόνο προγράμματα και δράσεις των οποίων το αποτέλεσμα πρέπει να είναι εκ των προτέρων μετρήσιμο, αλλά θα πρέπει εκ των υστέρων και σε πολλές περιπτώσεις να μετράμε το αποτέλεσμα. Και σε ό,τι αφορά λοιπόν το πρόγραμμα καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, δεν φτάνει να βάζουμε τους νέους σε μια θέση μαθητείας. Θα πρέπει να παρακολουθούμε και τι γίνεται για να δούμε κατά πόσο είναι οι προσπάθειές τους και οι προσπάθειές μας έχουν στεφτεί με επιτυχία ή όχι. Τέλος, Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των μισθών και το πόσο επηρεάζει αυτό την οικονομική ανάπτυξη είναι σαφές νομίζω για όλους. θέμα, είναι ένα θέμα που εξετάζουμε και στις συστάσεις κατά αναχώρα. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ισορροπία μεταξύ της εγχώριας ε, ζήτησης και της ανταγωνιστικότητας μιας χώρας. Για να δούμε και πώς εξελίσσεται η παραγωγικότητα σε επίπεδο κράτος μέλους. Αυτός είναι ο μύτος ο οποίος διατρέχει όλες τις εκθέσεις αυτές. Τι άλλο. Η κοινωνία των πολιτών. Και το κοινοβούλιο και οι κοινωνικοί εταιρεία θα πρέπει να συμμετέχουν πιο πολύ. Αλλά ναι, θα συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών. Προβλέπετε αυτό. Σας διαβεβαιώνω. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Τομπρόφσκη. Uh, ε, ε. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα επικεντρωθώ μάλλον σε δύο θέματα. Πρώτο, στην ερώτηση που έγινε όσον αφορά την ταχεία μείωση των ελλημάτων. Για να επαναλάβω απλά τα όσα προαναφέρθηκαν στις εισαγωγικές παρατηρήσεις, ότι ουσιαστικά εφέτος και του χρόνου 2015 αναμένουμε μια ουδέτερη δημοσιονομική κατάσταση. Ούτε επέκταση δημοσιονομική αναμένουμε, ούτε συνολική λιτότητα ή πειθαρχία εξετάζοντας φυσικά όλες τις χώρες ε, ε, συνολικά από κοινού. Υπάρχουν όμως κάποιες χώρες που υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα όσον αφορά τα ελλείμματα εκεί και περισσότερες προσπάθειες πρέπει να γίνουν. Αλλά γενικά αναμένουμε μια ουδέτερη δημοσιονομική κατάσταση και αυτό είναι κάτι το σημαντικό όσον αφορά τις εξελίξεις. Και δεύτερον, αναμένουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα από το 2,6% του ΑΕΠ να μειωθεί σε 2,4% του ΑΕΠ. Και αυτό θα συμβεί όχι μόνο λόγω της ε, ε, λιτότητας όσον αφορά την εξέλιξη του ΑΕΠ αλλά και λόγω της οικονομικής ανάπτυξης συνολικά. Σίγουρα λοιπόν υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Και επίσης θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Βάνα όσον αφορά την εμπλοκή και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και όσον αφορά και τον κοινωνικό διάλογο με τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι κάτι επί του οποίου εργαζόμαστε τώρα στην προσπάθεια ένταξης αυτών των στοιχείων στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να ενδυναμώσουμε επίσης ε, την, ε, τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και επίσης ε, και κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ε, πράγμα που αναδείχθηκε, την ενδυνάμωση του ρόλου των ε, Ευρωπαίων εταίρων σε σχέση με τα στοιχεία της ετήσιας ε, επισκόπησης και την ενδυνάμωση των προτεραιοτήτων ε, των ε, εταίρων σε σχέση με συγκεκριμένες συστάσεις. Προτείνουμε κάποιες προσαρμογές λοιπόν όσο αφορά το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για να επιτραπεί καλύτερη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους αλλά επίσης και με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τα κοινοβούλια, ευρωπαϊκά κοινοβούλια των κρατών μελών. Αυτό είναι ακριβώς αυτό το οποίο πράττουμε αυτή τη στιγμή. Σε αυτό επικεντρωνόμαστε. Να δούμε πώς θα εργαστούμε ώστε να βελτιωθεί σφαιρικά, συνολικά η εμπλοκή των διαφόρων ε, συνεισφερόντων και εμπλεκόμενων όσον αφορά την ε, τον πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει να έχουν σε αυτές τις διεργασίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επίτροπε Μοσκοβισή, παρακαλώ. Για τον τελευταίο λόγο. Ναι, για να πατήσω. Δεν πιστεύω, το είχα πει και στην ακρόασή μου, ότι η κρίση ε, δεν ήταν σε βαθιά κρίση. Ε, έχουμε αρχίσει μια πολύ ισχνή ανάπτυξη και αυτή τη στιγμή έχουμε ε, υπό ανάπτυξη, υπό και φυσικά πολύ μεγάλη ανεργία και αυτό οδήγησε σε μια κοινωνική και πολιτική κρίση. Ε, γι' αυτό και ο πρόεδρος ε, Γιούγκερ θεωρεί ότι η Επιτροπή αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο η Επιτροπή της τελευταίας ευκαιρίας. Ε, δεν είναι αυτό που πιστεύω, ε, κυρία μου, πραγματικά. Αυτό που πιστεύω και ε, το δήλωσα και το υποστηρίζω είναι ότι το γεγονός ότι έχουμε περιέλθει σε αυτή την κατάσταση δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να κάνουμε δημοσιονομική εξηγίαση, μείωση των ελλημάτων, και να υπάρχει μείωση όλων αυτών των δαπανών. Όπως είπε και ο κύριος Ντομπρόσκη, το έλλειμμα εξακολουθεί να μειώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημοσιονομική πειθαρχία θα επιβραδυνθεί για πολλές χώρες ε, για τον απλό ούστατο λόγο ότι έκαναν τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε και αυτοί που δεν το έκαναν θα πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν. Και αυτή είναι η απόφαση που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Παρασκευή ε, προχθές. Αλλά πέραν αυτού θα ήθελα να προσθέσω το εξής το είπα και το ξαναλέω εδώ, ότι οι κανόνες όσοι έχουν δεν είναι φλακώδεις σε καμία περίπτωση, επιτρέπουν ένα περιθώριο ευελιξία το οποίο σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε και να ε, χρησιμοποιήσουμε στην Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή και θα υπάρχει και στην ανακοίνωση που σας είπε ο Βαλτής ε, στις αρχές Ιανουαρίου για να σας πούμε ποιες είναι οι ευελιξίες και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι ευελιξίες στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και επίσης να σας πω ότι υπήρχε και μια διάσταση η οποία δεν υπήρχε στην παρούσα οικονομική πολιτική μέχρι τώρα και που σχετιζόταν σίγουρα και με το έλλειμμα αντίληψης είναι η διάσταση των επενδύσεων. Οι επενδύσεις είναι αυτές οι οποίες ακριβώς τιμωρούν σε μεγάλο βαθμό την Ευρώπη σε σχέση με τους μεγάλους ανταγωνιστές της και γι' αυτό ακριβώς και το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε την περασμένη Τετάρτη προσπαθεί να επανορθώσει την κατάσταση. Ευχαριστώ όλους. Ζητώ συγγνώμη, διότι 10 άτομα επιπλέον ήθελαν να θέσουν ερώτηση και δεν υπήρχε αρκετό χρόνο. Είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες συναντήσεις και θα υπάρχει δυνατότητα να τεθούν ερωτήσεις και να ληφθούν απαντήσεις από τους τρεις επιτρόπους. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά σας. Και όπως είπε και ο Επίτροπος Μοσκοβισή, ναι μεν έχουμε ακόμα κρίση, αλλά υπάρχουν ελπίδες και δυνατότητες ε, μπροστά μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Well, I have to leave this... Εγώ πρέπει να αποχωρήσω γιατί έχω μία ακρόαση για το TTIP σε άλλη συνεδρίαση. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Δέκα άτομα από εσά δεν μπόρεσαν να λάβουν το λόγο, αλλά εσείς δεν ήσασταν στον κατάλογο των αγορητών. Ευχαριστώ.